φυσικά καλό τους πάντες να στηρίξουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Αρής. Έληξε και σας υπενθυμίζω και εγώ από την πλευρά μου την ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Ρης θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτήρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του διαδικτύου πρόγραμμα NSA PRISM. Θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για τη συζήτηση αυτή θα υπάρξει ένας γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και ότι δεν προβλέπεται διαδικασία catch the eye, ούτε γίνονται δεκτές οι μπλε κάρτες. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής στον Επίτροπο Μπόρτς για τα εισαγωγικά του σχόλια. Commissioner Ναι, κυρία Πρόεδρε. Θα διαβάσω τη δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής. Αντικαθιστώ την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ που δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για πρόσφατες ανακοινώσεις των μέσων ενημέρωση ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται σε ευρεία βάση τα στοιχεία των ευρωπαϊκών πολιτών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες online. Προγράμματα όπως το πρόγραμμα PRISM και η βάση των οποίων εφαρμόζονται και επιτρέπονται αυτά τα προγράμματα αποτελούν κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η περίπτωση αυτή που αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης πιθανότατα να ενισχύσει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τη χρήση των ιδιωτικών στοιχείων τους ε, online και στο cloud. Το 2012, 70% των Ευρωπαίων πολιτών ανησυχούσαν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους είχαν συγκεντρωθεί η περίπτωση πίσω που αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζει τις διαφορές ανάμεσα στην, Ευρωπαϊκή, ε, στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ στο θέμα της προστασίας των δεδομένων. Ενώ στις ΗΠΑ το νομικό, νομοθετικό σύστημα προβλέπει ότι μόνο οι Αμερικανοί πολίτες και κάτοικοι προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα όλα τα προσωπικά δεδομένα και η εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους αναγνωρίζονται και προστατεύονται ως θεμελιώδη δικαιώματα ανεξάρτητα από την εθνικότητα του ατόμου ενώ εκθέσεις, ε, οι πληροφορίες που δεχόμαστε είναι ανησυχητικέ, το νομικό θέμα δεν είναι κάτι το καινούριο. Αντιμετωπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο παρελθόν. Για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, η Επιτροπή έχει θέσει το θέμα της, εφαρμογής, της υπερβολικής εφαρμογής του νόμου σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο των συνεχιζομένων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε για μια συμφωνία γενική προστασίας δεδομένων σε ό,τι αφορά την αστυνομία και την, νομική, και την δικαστική συνεργασία. Η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ έχει λάβει εντολή να διαπραγματευτεί αυτή τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε και θα ενημερώνει τα μέλη και ειδικότερα τα μέλη της ομικής Επιτροπής για τις εξελίξεις αυτών των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή ζητά σαφέστερη ε, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ε, ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων τους και σε, σε δικαστικά μέσα, σε δικαστικές λύσεις, έτσι όπως προβλέπεται για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα PRISM, η Επιτροπή θα θέσει το θέμα αυτό, πρίσμα, θα θέσει το θέμα αυτό με τις Ηνωμένε Πολιτείε με την πρώτη ευκαιρία. Θα ζητήσει διευκρινήσεις σε ο, για, το κατά πόσο πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια του προγράμματο PRISM περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και βασίζεται σε συγκεκριμένες υποψίες ή επιτρέπει την μαζική μεταβίβαση δεδομένων. Η αντιπρόεδρος κύριος Ρέντινγκ θα θέσει το θέμα με έμφαση και αποφασιστικότητα στην επικείμενη ε, Υπουργική Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, Ηνωμένων Πολιτειών στο Δουβλίνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενεργήσει επίσης εξασφαλίζοντας ότι θα ευωδιαστεί με την κατάλληλη νομοθεσία που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες καταστάσεις και αναφέρομαι ειδικότερα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την τρέχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οδηγία για την προστασία των δεδομένων, όταν τα δικαιώματα ενός πολίτη σε κράτος μέλος ε, ε, ε, αντιμετωπίζονται θα αποφασίσει ο δικαστής κατά φόσον πρέπει να μεταφερθούν νόμιμα τα δεδομένα σύμφωνα με τις δικαστικές ε, απαιτήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ευρύτερα. Αυτό είναι και ο σκοπός της ε, του προτινόμενου κανονισμού για τη γενική προστασία δεδομένων. Η έκθεση της κυρίας ε, της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ διατηρεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επικυροποιώντας τα δικαιώματα των πολιτών και εξασφαλίζοντας ε, την ενημέρωσή τους για την τυχόν καταπάτηση των δικαιωμάτων τους και όταν απαιτείται η έγκρισή τους, η έγκριση αυτή να είναι ουσιαστική. Πιο συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκή των, της προστασίας των δεδομένων πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κατά, προβλήματα όπως το πρόγραμμα PRISM μέσα από τους δικούς της κανόνες και τις δικές της διατάξεις σε για να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό έδαφος. Όταν εταιρείες, υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα στους Ευρωπαίους καταναλωτές θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τον Ευρωπαϊκό Νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να υπάρχει ευθύνη για εκείνους ε, που επεξεργάζονται τα δεδομένα και επίσης για εκείνους που μεταφέρουν, μεταφέρουν και μεταβιβάζουν προσωπικά δεδομένα. Η άποψή μας είναι ότι για να αποφύγουμε σύγκρουση δικαιοδοσίας η πρόσβαση σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές με αποτέλεσμα την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ε, Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στους servers αμερικανικών εταιριών πρέπει να καλύπτονται από συγκεκριμένους κανόνες στο πλαίσιο των συμφωνιών αμοιβαίας παροχής ε, υπηρεσιών που ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί περισσότερο στη διατάξη του κανονισμού οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η απόφαση ενός δικαστηρίου τρίτης χώρας μπορεί να εφαρμοστεί ε, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει αυτές τις προτάσεις. Αξιότιμα μέλη, κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή πιστεύει ότι η γρήγορη ε, υιοθέτηση αυτής της πρότασης θα λύσει οποιαδήποτε νομικά κενά τα οποία δημιουργούνται όταν εταιρείες συλλέγουν και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών και που υπόκεινται σε διαφορετικές κυριαρχίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τους στόχους και τις αρχές της μεταρρύθμισης της προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων και να προβεί στην ταχύτατη έγκριση αυτού του πακέτου. Σα ευχαριστώ πολύ, Πίτρο Περπόρτ, Και τώρα οι μιλητέ από τι πολιτικέ ομάδε και καταρχήν ο κύριο Βέμπερ, εξ ονόματο του ΕΛΚΑ, για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, τα δεδομένα μου μου ανήκουν. Αυτή αυτό είναι το οδηγό νήμα της ευρωπαϊκής σκέψης και το κράτος βασίζεται σε αυτή την αρχή ότι τα δεδομένα του πολίτη ανήκουν στον πολίτη. Αυτή λοιπόν είναι μια αρχή την οποία πρέπει να σέβονται όλα τα κράτη και το κράτος καλείται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις κόκκινες γραμμές. Γι' αυτό λοιπόν οι εκτάσεις από τις ΗΠΑ είναι ανησυχητικές, είναι πάρα πολύ καλό που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και είναι πολύ σωστό το ότι ξεκινάει μια νέα διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ευαισθητοποίηση για προσωπικά δεδομένα. Είναι απαράδεκτο λοιπόν και αυτό το εκφράζω εκ μέρους του ΕΛΚ το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, διαφοροποιούν τα δεδομένα κατά πόσον αφορούν αλλοδαπούς ή μεδαπούς. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι Αμερικανοί φίλοι μας. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση μπροστά μας και πρέπει να ορίσουμε τους στόχους μας. Πρώτον, χρειαζόμαστε διαφάνεια, να ξέρουμε τι θα συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή, κυρίως η Αντιπρόεδρος ε, κυρία Ρέντινγκ, χέρι της πλήρους ε, και αμέριστη υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συζητή στο εκεί όπου θα τεθούν αποτελούν επιτάπητος η νομική βάση και η εφαρμογή μέτρων. Δεύτερον, θέλουμε διαφάνεια όσον αφορά τι εταιρείε. Google, Facebook, αυτοί κερδίζουν πολλά χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτε λοιπόν, άρα οι πελάτε αυτών των εταιριών, έχουν δικαίωμα σε διαφάνεια. Μήπω έχουν αυτόματη πρόσβαση σε δεδομένα ή όχι. Τρίτον, θέλουμε να διευκρινίσουμε το ρόλο τη ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν πληροφορίε ότι αυτοί έχουν ειδική πρόσβαση στα δεδομένα των Ευρωπαϊκών Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει η Βρετανική κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Τέταρτον, το ίντερνετ είναι παγκόσμιο, γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινέ προδιαγραφέ. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν επεξεργάζεται ένα νόμο πλαίσιο που αφορά την ε, αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Καλό αυτό, αλλά ε, δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε ε, συνεργασία μόνο σε αστυνομική ε, φύσεως θέματα, αλλά συνεργασία και σε θέματα δεδομένων. Ένα τέτοιου είδους, ε, μια τέτοιου είδους συμφωνία πλαίσιο χρειαζόμαστε. Κατόπιν, χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό cloud. Όταν αποθηκεύονται δεδομένα στο ευρωπαϊκό cloud, να αποθηκεύονται στην Ευρώπη, γιατί μόνο τότε οι εταιρείε μπορούν να μας εγγυηθούν ότι ε, για τα δεδομένα αυτά ισχύουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και έκτον, χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο δίκαιο περί ε, δεδομένων γιατί μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε στους Αμερικανούς κοιτάξτε εμείς στην Ευρώπη έχουμε σύγχρονες προδιαγραφές και θέλω επίσης να πω ότι κάποιες εξελίξεις στον τομέα αυτό με ανησυχούν διότι σωρεύονται δεδομένα υπάρχουν και δυνατότητες ε, εκμετάλλευσης αυτών των δεδομένων άρα δηλαδή σήμερα πρέπει να έχουμε το θάρρος να τραβάμε κόκκινες γραμμές όπως το προτείνει η Κομισιόν και θέλω να πω ε, στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μην ξεχνάτε, στις 9 Ιουλίου θα ψηφίσουμε. Να μην μας κατηγορήσουν ότι εμείς καθυστερούμε. Και απευθύνουμε στο Συμβούλιο. Ας πάψετε πια να αναφέρεστε σε αμεληταία θέματα, σε λεπτομέρειες, να αντιμετωπίσετε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής. Και τελευταίο σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, για το ΕΛΚ είναι πολύ σημαντικό να πούμε το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι συνεργάτες μας. Το PNR, στο SWIFT, εμείς ως Ευρωπαίοι δεν μπορέσαμε να παρουσιάσουμε προδιαγραφές. Ε, και όσον αφορά το, την εγκληματικότητα, το, την τρομοκρατία, δεν μπορέσαμε να την αναχαιτήσουμε. Όμως οι Ευρωπαίοι επωφεληθήκαμε. Ας πούμε στη Γερμανία προλάβαμε την ε, ε, αποτροπή ε, μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Το ίδιο συνέβη και στη Μαδρίτη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σε επισημάνω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι συνεργάτες μας. Ειδικά για το SWIFT περιμένουμε την αξιολόγηση των δεδομένων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής κατά πόσον το SWIFT μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις ε, ε, μεταφορές ε, κονδυλίων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, εφόσον οι ΗΠΑ είναι συνεργάτες μας, από κοινού καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, και τώρα ο κύριος Μωράης, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ε, Πέτροπε, για τους σοσιαλιστές τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα Guardian την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με το σύστημα που αποκαλείται Prisma και το οποίο διαχειρίζεται η NSA, που οδηθεύεται σε συνεργασία με γίγαντες της πληροφορικής όπως η Apple, Google, Microsoft, Skype, YouTube και οι μεγάλες γιγάντιες εταιρείες ε, για την κατασκοπία έχουν προκαλέσει τεράστιες ανησυχίες στις, ε, στις, στους πολίτες μας έχει υπάρξει μια τεράστια, ένα τεράστιο ε, ρήξη εμπιστοσύνη και για μα η Υπουργική Συνεδρίαση 13 και 14 Ιουνίου είναι κάτι που θεωρούμε ζωτική σημασία. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει, καθώ και όλε οι πολιτικέ ομάδε, να στηρίξουν τον Επίτροπο και να ε, και να θεωρήσουν υπόλογες της ΕΠΑ για αυτό που έκαναν, για τη μεταφορά δηλαδή προσωπικών πληροφοριών των πολιτών μας που μπορεί και τελείως να είναι περιττό στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και στην υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών μας. Σε περιττές πληροφορίες που απλώς ε, ε, μειώνουν την εμπιστοσύνη και όλα αυτά υποτίθεται στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάγκη προστασία δεδομένων. Αυτή, αυτή είναι πολύ σημαντική ισορροπία. Η έκθεση στην Guardian και στην ε, Washington Post της Νέας Υόρκης ε, σημαίνει, δείχνει ότι αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούν ε, αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με συγκεκριμένες δικαστικές εντολές και τους δίνεται, δίνεται πρόσβαση στους σερβερς τους για τις Αμερικανικές αρχές. Υπάρχει μάλιστα δυνατότητα να στέλνονται άμεσα στις εταιρείες που χειρίζονται αυτά τα στοιχεία. Επίσης ανησυχητική είναι η γενικευμένη πρόσβαση στα, ευρωπαϊκά, στα στοιχεία Ευρωπαίων πολιτών και μπορεί και αυτό να έχει γίνει υπό την ευθύνη των ε, προαναφερθήσεων εταιριών. Δεν υπάρχει συμμόρφωση με την ε, ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης ανησυχούμε για την απουσία ενός γενικού υπερατλαντικού νομικού πλαισίου για την εξασφάλιση της προστασίας των στοιχείων. Επίσης δεδομένου ότι υπάρχει διαπραγμάτευση Συνεχίζονται από το 2011 διαπραγματεύσεις σε σχέση με την ε, ανταλλαγή στοιχείων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλους αυτούς τους λόγους θα θέλαμε ο Επίτροπος ε, να ζητήσει λογαριασμό από τη ΣΥΠΑ και να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές των ΗΠΑ όταν επεξεργάζονται ε, στοιχεία αλλοδαπών πολιτών να το κάνουν με τα δικά μας ε, πρότυπα. Επίσης θέλουμε να δεσμευτείτε για μια συμφωνία υψηλού επίπεδου για το πακέτο προστασίας των δεδομένων με βάση τις γραμμές που έχουμε εμείς υποβάλει ε, με των εισηγητών μας και των σκιωδών μας όσον αφορά την αύξηση της προστασίας των δεδομένων. Θα πρέπει να προστατεύονται η χρήση των στοιχείων δεν μπορεί να καθυστερήσει πλέον μια τέτοια νομοθεσία. Επίσης, σε θέματα που αφορούν την ε, προστασία των δεδομένων θα ε, συζητηθούν ε, κατά τη διάρκεια όλων των συμφωνιών με τη ΣΥΠΑ ώστε να διατηρηθεί η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γνωρίζουμε την πρόθεση της Κομισιόν να ζητήσει λογαριασμό από τη ΣΥΠΑ σε σχέση με τις ροές πληροστοιχείων, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό το φως του πρίσμα και του NSA και της υπόθεσης οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι βέβαιοι για το τι μπορεί να συμβεί. Στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν πολύ σοβαρές ανησυχίες για το τι συνέβη και θεωρούν ότι αυτή η ρήξη, αυτή η παραβίαση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη, να φροντίσει ώστε να διατηρηθούν οι δικές μας προδιαγραφές και ότι θα προστατευτούν οι Ευρωπαίοι πολίτε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μωράης, να σας θυμίσω συνάδελφοι ότι σύμφωνα με την απόφαση των πολιτικών ομάδων δεν υπάρχει διαδικασία κάτσε διάει εδώ, ούτε μπλε κάρτες επιτρέπονται σε αυτή τη συζήτηση και αυτό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνο για τους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω την, από τη συνάδελφο Ιντεφέλτ εξ ονόματος των Φιλελευθέρων για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε ένα τεράστιο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών σοκαρίστηκαν ότι ένα ξένο κράτο έχει απεριόριστη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία της ζωής τους. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θεωρείται αυτό σε όπω όπως λένε οι Γερμανοί. Και ο ίδιος ο πρόεδρος απάντησε σε ερωτήματα του Κογκρέσου και των μέσων ενημέρωσης για αυτό το θέμα τι, αυτά που, τι ε, συμβαίνει στην Ευρώπη. Με όλο το σεβασμό που οφείλω στον Επίτροπο, ο Επίτροπος Δημόσιας Υγείας έρχεται εδώ για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ενώ ο Πρόεδρος Μπαρόσο θα έπρεπε να είχε πάρει το ελικόπτερό του και να έρθει τρέχοντας στο Στρασβούργο για να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών. Έχουμε τουλάχιστον έναν υπεύθυνο για τον Επίτροπο για την Αντιμοκρατία στο Κοινοβούλιο. Πού είναι αυτός. Γιατί δεν είναι εδώ οι πολιτικοί ηγέτε τη Ευρώπη, Αλλά πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει με εμά, συνάδελφοι. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το μισοάδιο ε, ημικύκλιο. Ενώ αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα είχαμε στο παρελθόν αποφασίσει να δημιουργήσουμε μία ομάδα ε, μελέτης για το έσλον. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δεν ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε και να κάνουμε κάτι. Δεν, μπορούμε να... δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι μας παρακολουθούν ακολουθούν οι Αμερικανοί. Το ξέραμε αυτό. Έχουμε υποβάλει τα σχετικά ερωτήματα κατά επανάληψη. Αλλά το να υποβάλουμε ερωτήματα στην Επιτροπή είναι σαν να μιλάμε σε, με ένα τείχο. Έχω ένα μακρύ κατάλογο μη απαντήσεων στα ερωτήματα που είχα υποβάλει για, το, για ένα σωρό θέματα ε, και, σημεία του Αμερικανικού δικαίου χωρίς να πάρουμε ποτέ απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη, επειδή γίνεται μια εθνική συζήτηση παντού για αυτό το θέμα, η κυρία Μέρκελ θα ζητήσει, ε, θα ζητήσει εξηγήσει από τους Αμερικανούς. Όλα τα κράτη-μέλη ε, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου και εκείνου του κυρίου Μόρε στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνουν το ίδιο. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες. Δεν το κάνουμε και γι' αυτό χάνουμε την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις τους, αλλά ούτε και οι κυβερνήσεις έχουν εμπιστοσύνη στους πολίτες τους. Χάνουμε ηθικό ε, βάρος εδώ. Πώς μπορούμε να πούμε, τι θα πούμε σε μια χώρα όπως την, Αίγυ, ε, την Αίγυπτο, το Ιράν, πώς μπορούμε να τους πούμε ότι δεν πρέπει να ε, παρακολουθείτε τους πολίτες σας, διότι αυτό είναι αντιδημοκρατικό, όταν κάνουμε εμείς το ίδιο για τους δικούς μας πολίτες. Χάνουμε την αξιοπιστία μας εδώ και σε ό,τι αφορά την ειδική σχέση άκουσα όλους τους συναδέλφους να αναφέρονται στην ειδική σχέση με τους καλύτερους φίλους και τους πλησιέστερους συμμάχους μας που είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη δήλωση του Προέδρου Ομπάμα όταν απευθυνόταν σε ένα Αμερικανικό ακροατήριο που ανησυχούσε. Τους είπε μην ανησυχείτε, δεν παρακολουθούμε εσά τους ε, Αμερικανούς πολίτες, παρακολουθούμε τους ξένους. Οι ξένοι είμαστε εμείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί λοιπόν ειδική σχέση μιλάμε. Επί 12 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι η πλησιέστερη σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της ομοκρατίας. Θα παραμείνουμε τέτοιοι σύμμαχοι. Αλλά χρειαζόμαστε ίση αντιμετώπιση. Απευθύνομαι, απευθύνομαι ε, στον Επίτροπο λέγοντας ότι αυτό είναι σεφζάχ, σημαντικό θέμα που πρέπει να αναλυφθεί από πολιτική ηγεσία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και τώρα εκ μέρους των ε, Πρεσιών συνάδελφος κύριος ε, Albrecht. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά Επίτροπε. Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που ελέγχθησαν από τις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για την προστασία δεδομένων, δεν διακυβεύεται ένα αμεληταίο τεχνικό θέμα, διακυβεύεται το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με μαζική παρακολούθηση πολιτών ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα δηλαδή πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε μαζική παρακολούθηση. Χρειαζόμαστε ισχυρούς ε, κανόνες για την προστασία δεδομένων, για τη στήριξη της δημοκρατίας δημοκρατίας, του κράτου δικαίου, τη ασφάλεια, τη εμπιστοσύνη, στην αγορά, την ψηφιακή αγορά και γενικότερα την αγορά στο σύνολό τη. Άρα δηλαδή πρέπει να αντιδράσουμε ω Ευρωπαίοι, να συστήσουμε τι δικέ μα τι προδιαγραφέ για την προστασία των δεδομένων, να διαφυλάσσουμε καταρχήν τα δικαιώματα των δικών μα των πολιτών και να αποφασίσουμε το συντομότερο δυνατόν επί τη προτινόμενη νομολογία και νομοθεσία, γιατί σε τελική ανάλυση εδώ ε, πρόκειται για όγκους δεδομένων για μαζική παρακολούθηση. Εάν λοιπόν πραγματικά επιθυμούμε να έχουμε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό cloud, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων που θα μπορούν να εφαρμόζονται και που θα δημιουργούν ε, και μία σαφήνεια για τη μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες. Ως ε, ε, συγητής της Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων με τις ΗΠΑ θέλω να πω ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε προδιαγραφές, αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και κάποιες κινήσεις. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές, γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινή βάση συζήτησης. Στον συνάδελφο Κικ από το ECR για τρία λεπτά. Uh, President, uh, Commissioner. Πρόεδρε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση αφορά την αύξηση της εμπιστοσύνης ε, και της πίστης των πολιτών, καθώς και να ε, εξηγηθούν κυβερνήσεις και υπηρεσίες που τους υπηρετούν και τους προστατεύουν. Αυτές οι εταιρείε που ήδη έχουν κατονομαστεί έχουν αρνηθεί ότι έχουν ενεργήσει παράνομα. Οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασαν την ε, ανησυχία τους, τα ακούσαμε και σήμερα το πρωί, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι αυτή τη στιγμή πολύ νωρίς για να καταλήξουμε συμπεράσματα. Ωστόσο, ήδη εμείς ε, δαχτυλοδείχνουμε και ορισμένοι ε, εκφράζουν ε, αντιαμερικανικές ρήσεις όπου είναι πολύ οικίες όπως είναι και ο τυχοδιοκτισμός και η μεγαλοστομία χωρίς αποδείξεις δεν μπορεί κανείς να καταδικάζει έναν κατηγορούμενο πριν να γίνει δίκη. Το Κοινοβούλιο εργάζεται πολύ, συχνά, πολύ σκληρά μάλλον για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και για την ανταλλαγή υπόρου των στοιχείων, κάτι το οποίο ε, υποστηρίζουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας πέρα από τα σύνορά μας ε, μέσω των σχέσεων μας με άλλες χώρες. Και ήθελα να σας προειδοποιήσω γιατί συχνά κάποιοι ευρωβουλευτές δείχνουν ότι πολύ λίγα μας ενώνουν ε, στις αξίες, ε, αντίθετα μας απομακρύνουν. Η προστασία των πολιτών από σύγχρονες απειλές είναι ένα ε, έργο δύσκολο και πολύ συχνά υπάρχει, μάλλον κατηγορούνται οι αρμόδιοι ότι δεν προχωρούν αρκετά ενώ από την άλλη μπορεί να κατηγορηθούν ότι προχώρησαν υπερβολικά πολύ. Ε, όλο ένα και περισσότερο οι τρομοκράτες και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν την ε, τεχνολογία της πληροφορίας κατά των πολιτών μας. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προσδοκίες ώστε η ίδια η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί προς όφελόν μας. Αυτές οι πληροφορίες φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πλαίσια δημοκρατικών αρχών και νομικής εποπτείας. Ωστόσο, δεν, πρέπει να κατανοήσουμε, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι κερδίζουμε περισσότερες ελευθερίες όταν αφαιρούμε ελευθερίες άλλων και ότι το κυριότερο είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Γι' αυτό και είναι πιο σημαντικό για μας τους πολιτικούς που να θυμίζουμε ότι η εξασφάλιση της ασφάλειας και της ελευθερίας των συμπολιτών μας δεν θα πρέπει να ε, την εγγυόμαστε με την ε, θυσία της δημοκρατίας. Ωστόσο θα πρέπει να θυμίζουμε και ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός και που βρίσκεται. Και όταν έχουμε να κάνουμε με τους συμμάχους μας και θέλουμε απαντήσεις και την αλήθεια, οι φίλοι είναι αυτοί που ακούν περισσότερο όταν μιλάς και όχι όταν ουρλιάζεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Πάσκα, εξ του EFT, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, με φοβερά αυτές οι διαρροές του προγράμματος PRISM. Η, υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία συγκεντρώνει στοιχεία, αξιολογεί τα στοιχεία για τους πολίτες μας. Αξιολογεί όλες τις επικοινωνίες που γίνονται μέσω αμερικανικών καναλιών. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάζουν την ιδιωτικό βίο, την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την παράνομη παρακολούθηση ε, των ε, πολιτών μας από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Γι' αυτό οι αμερικανικές εταιρείες που έχουν πρόσβαση, επιτρέψει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε, να ρεδιευνήσουμε και να εφαρμόσουμε τα ίδια μέτρα και τις ίδιες κυρώσεις που ισχύουν για άλλους οι οποίοι παραβιάζουν τους νόμους μας. Η παρανοϊκή συμπεριφορά των Αμερικανών εταίρων μας είναι πραγματικά θλιβερή. Και τώρα το λόγο έχει ε, συνάδελφος η κυρία Βερζιά, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούγοντα σας κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας πω, μήπως μας κοροϊδεύετε, δεν γνωρίζετε τίποτε για το θέμα. Θα πρέπει να είναι παρούσα εδώ η κυρία Ρέντιν και θα ήθελα να πω, υπάρχει κάτι το νέο υπό τον ήλιο, ε, τον υπερατλαντικό ήλιο. Αυτά που ακούσαμε επιβεβαιώνουν ότι μόνο λίγοι από εμάς, κάτι που καταγγέλουν διαρκώς, ενώ μιλάμε για την προστασία, προστασία των προσωπικών δεδομένων θυμάμαι τον Ντένις το 2010 να μας λέει πώς η ιδιωτική ζωή των Αμερικανών ε, πολιτών προστατεύεται από την Αμερικανική νομοθεσία. Ο ρυθμός εκείνων που αφιβάλλουν αυξήθηκε ε, πρόσφατα. Χάρη στον Γουάντεν γνωρίζουμε ότι η NSA έχει άμεση πρόσβαση στα, ε, στους σερβέρς των μεγάλων, των μεγάλων εταιριών ίντερνετ. Οι απαντήσεις είναι Μα δεν είχαμε ιδέα. Θα εξετάσουμε όλα τα αιτήματα με προσωπική. Το σημαντικό για εμά του Ευρωπαίους κάτι που βγήκε από το στόμα, είναι κάτι που βγήκε από το στόμα του Προέδρου Ομπάμα. Δεν ήταν οξεμολόγηση, διότι είπε βάση δικαίου η παραγωγή του Ιντερνετ δεν ισχύει για τους Αμερικανούς υπηκόους ή τους Αμερικανούς κατοίκους. Η κατασκευη το να επιτρέπεται να κατασκοπεύονται οι κινήσεις των Αμερικανών πολιτών, αλλά φαίνεται δυστυχώς ότι αυτό γίνεται και για τους πολίτες άλλων χωρών. Και αυτό το υπογραμμίζουμε εδώ και χρόνια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που ισχύουν για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεντρώνονται στοιχεία σε, μεγάλο όγκο ε, ε, ε, οι υπηρεσίες ελέγχου του... της Europol μας το υπογραμμίζουν αυτό διαρκώς. Επιτέλους λοιπόν δεν, δεν μπορούμε πλέον να δεχόμαστε να έρχονται οι απεσταλμένοι σας και να μην έχουν τίποτε να μας πούν. Απορρίψαμε την άκτα επειδή θέλαμε οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Παρακράτησε αυτό. Τέρμα υποκρισία έχουμε υπερβολικά πολλά στοιχεία για, το, για αυτά που λέμε και για αυτά που ισχυριζόμαστε. Πρέπει να απαιτήσουμε από τους Αμερικανούς, από την, Αμερικανική, ε, από την Αμερική την προστασία των, πολιτών, δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Τελ. Άουζερ από τους μη γεγραμμένους για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα λέγατε εάν ε, μια μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ε, σας παρακολουθούσε κύριε Επίτροπε ολόκληρο το 24ωρο φαντάζομαι δεν θα συμφωνούσατε έτσι δεν είναι αλλά κοιτάξτε ακριβώς αυτό συμβαίνει στον ψηφιακό χώρο 24 ώρες ε, της ημέρας παρακολουθούνται εκατομμύρια ανθρώπων και εδώ εμείς είμαστε αρμόδιοι για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων το πρόγραμμα που τρέχει παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα και τι κάνουμε εμείς εμείς λέμε τόσο στο SWIFT, όσο και ο PNR, ότι εντάξει θα δεχτούμε αυτά που λένε οι Αμερικανοί. Δεν γίνεται όμως αυτό. Επιτέλους πρέπει να αναλάβουμε εμεί τα ενία, να αναλάβουμε τις ευθύνε μας, να ασκήσουμε πίεση, έτσι ώστε να ανακληθεί αυτό το πρόγραμμα και να δρομολογήσουμε και έρευνες για να δούμε τις νομικές προεκτάσεις αυτού του προγράμματος. Ποιος επωφελείται από αυτό το πρόγραμμα, μήπως επωφελείται η Europol. Και σε τελική ανάλυση ας έρθουν εδώ Αμερικανοί σε αυτό το χώρο ε, να ε, μας αποδώσουν λογαριασμό. Γιατί αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή απλά είναι μια παρέκκληση από την ελεύθερη δημοκρατία. Uh, Και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Μπόρτζ για τις ε, τελικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν θα πρέπει να πω ότι συμμερίζεται την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το σκάνδαλο πρίσμα και θα ενημερώσω την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ φυσικά για τη σημερινή μας συζήτηση. Θα πρέπει επίσης να δηλώσω όπως η κυρία Ρέντινγκ θα έρθει στην Επιτροπή Λίμπε στις 19 του Ιουνίου που σημαίνει ότι όχι μόνο θα συζητήσει και θα αναφέρει το θέμα και τις εξελίξεις ε, που θα έχουν υπάρξει μέχρι τότε, αλλά θα αναφερθεί και στην Επιτροπή για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που αναμένεται να γίνουν στο Δουβλίνο την επόμενη Παρασκευή και φυσικά θα αναφέρει τις κοινέ μας ανησυχίες στην Υπουργική Διάσκεψη της επόμενης εβδομάδας, στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο και φυσικά στους αρμόδιους Αμερικανούς. Ε, εκπροσώπου. Αυτή η συζήτηση ήταν πάρα πολύ καλή, κυρία Πρόεδρε, αν και ήταν σύντομη. Και φυσικά υπήρχαν δύο γραμμέ σκέψης που δεν είναι αντιφατικέ μεταξύ του. Μια από αυτέ είναι ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα με τη ΣΥΠΑ και να καταστήσουμε σαφές ότι οποτεδήποτε ένας Ευρωπαίος πολίτης, ε, μάλλον πληροφορίε ενό Ευρωπαίου πολίτη, ε, χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες και ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο προστασίας των στοιχείων από πλευρά των ΗΠΑ, ιδιαίτερα αν διαβάσετε όπως είπε και ο κύριος Μωράες, αν διαβάσει κανείς τον Guardian, την εφημερίδα Guardian. Υπάρχει αναφορά σε σχέση, από τον πληροφοριοδότη σε σχέση με την ευκολία με την οποία μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ε, από το ίδιο το άτομο το οποίο έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Η κυβέρνηση ε, λέει έδωσε στον εαυτό της ε, αρμοδιότητες που δεν μπορεί να έχει. Δεν επιτρέπεται να έχει. Δεν υπάρχει καμία δημόσια εποπτεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι όπως εγώ ίδιος έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε περισσότερο από όσο ε, μπορούμε κανονικά. Δηλαδή, μπορούμε λοιπόν να θέσουμε ερωτήματα στην επόμενη Υπουργική Διάσκεψη για το πόσο έχει γίνει αυτό σε σχέση με Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα ε, εκτιμώ τις παρατηρήσεις του κυρίου Κέρχοπ. Ε, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι ο εχθρός. Όπως είπε και εκείνος. Και εγώ μπορώ να το σχολιάζω ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών για 10 χρόνια. Τι σημαίνει ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας χωρίς τη συλλογή ε, στοιχείων και κατασκοπή, χωρίς κατασκοπία. Αλλά ε, το πρόβλημα κάθε υπηρεσίας επιβολής του νόμου είναι που ότι ενώ οι τρομοκράτες και το οργανωμένο έγκλημα δεν τηρούν κανένα νόμο, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε δημοκρατικές χώρες που διέπονται από το νόμο δίκαιο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρά τα αγάντια του νόμου για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Και γι' αυτό το λόγο Εκτιμώ τα σχόλια των όσων ε, είπαν ε, ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Έχουμε λύσει σημαντικά θέματα και έχουμε κάνει σημαντικές έρευνες όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας μέσω της ε, κοινή χρήση πληροφοριών με αυτόν τον ιδιαίτερο εταίρο μας, αλλά κανένας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή την ειδική σχέση για να παρακάμπτει τον νόμο και τις διεθνείς τις ε, προδιαγραφές. Ε, πολύ λεπτό το θέμα να διατηρήσουμε δηλαδή αυτήν την συνεργασία. Αλλά επειδή υπάρχει ακριβώς συνεργασία, σημαίνει όχι μόνο περισσότερα δικαιώματα, αλλά και περισσότερες υποχρεώσεις. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις λοιπόν και κανείς δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και να έχουμε υπόψη μας τα όσα είπε ο κύριος Κέρχοπ. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Να θυμίσω επίσης ότι στο πλαίσιο της πρότασης για τη μεταρρύθμιση της ε, προστασίας των δεδομένων και εκτιμώ τα σχόλια των διαφόρων ευρωβουλευτών όσον αφορά τη σημασία υιοθέτηση αυτού του νέου πακέτου που προτείνει η κυρία Ρέντινγκ, η Κομισιόν κατέστησε σαφές ότι οι έξω εδαφικές εφαρμογές νόμων από τρίτες χώρες μπορεί να είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η μεταρρύθμιση θεσπίζει νομικές οδούς που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η Κομισιόν είναι έτοιμη λοιπόν να εξετάσει οποιασδήποτε βελτιώσει θεωρήσει απαραίτητε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ω προ αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού για ταχεία υιοθέτηση αυτού του πακέτου, που μάλιστα ορισμένα κράτη θέλουν να καθυστερήσει. Ενώ είναι κοινό συμφέρον μα να δουλέψουμε χέρι με χέρι για την υιοθέτηση αυτού του πακέτου εν ώψη αυτών των πρόσφατων εξελίξεων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπόρτζ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, Σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της συναδέλφου Κοστέλο, Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους ε, απόρους. Θα δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια και θα παραδώσω την έδρα στον συνάδελφο Μαρτίνες.